Okay, now we have to... Yeah. Okay, colleagues, if we can take our... Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι για να ξεκινήσουμε αυτή την ειδική συνεδρίαση, ανταλλαγή απόψεων με τους νέους από την εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Νεολαία για το ρόλο της εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, ένα τεράστιο ζήτημα και Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολιτικές δυσκολίε και προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κάποια πολύ καλά πράγματα. Έχουμε χώρε που καλωσορίζουν τους μετανάστες και εργάζονται σκληρά για να εντάξουν ανθρώπους που ουσιαστικά εγκαταλείπουν κάποιε εμπόλεμε ζώνες. Επίση γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίε. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που θα, θα καλωσορίσω του σημερινού προσκεκλημένου μας. Ε, δεύτερη ε, συνεδρίαση τη εκδήλωσης Ευρωπαϊκής Νολέας έλαβε χώρα στις 20-21 Μαΐου. Είχαμε 7.000 νέους ανθρώπους που συζήτησαν τις ιδέες τους που παρουσιάζονται σε 10 διαφορετικές επιτροπές στο Κοινοβούλιο. Όλοι οι βουλευτές έχουν λάβει αντίγραφο της έκθεσης της εκδήλωσης για την Ευρωπαϊκή Νεολαία του Μαΐου, το Σεπτέμβριο. Το έγγραφο φέρει τον τίτλο «Διαμορφώνοντας στην Ευρώπη, 50 ιδέες για το μέλλον». Σήμερα έχουμε τρεις ομιλητές από την εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ελέα που θα μας παρουσιάσουν κάποιες ιδέες και κατόπιν θα σα ζητήσω να απαντήσετε στις ιδέες. Θα ακούσουμε, θα έχουμε λοιπόν τρεις σύντομε παρεμβάσεις από τους βουλευτές ιδίως θα είναι σύντομες οι παρεμβάσεις. Θα δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους μας, θα ακούσουμε τις ιδέες και θέλουμε τις δικές σα αντιδράσεις σε αυτές τις τρεις ιδέες δύο λεπτά για κάθε παρέμβαση το πολύ. Και ελπίζουμε ότι οι ιδέες που θα ακούσουμε από τους ε, καλεσμένους μας σήμερα θα τροφοδοτήσουν την επόμενη συνάντηση για την κοινή έκθεση μεταξύ ε, Επιτροπής ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ για τη μετανάστευση. Έχουμε τρεις ομιλητές. Λίδα Σλαπακόβα, οποία είναι αρμόδια διεθνών σχέσεων, ε, είναι εμπειρογνώμονα σε ευρωπαϊκές σπουδές ασφάλειας και ειρήνης και ασχολείται πιο συγκεκριμένα με το θέμα του εξτρεμισμού στην πολιτική ευρωπαϊκή Γειτονία. Έχει εργαστεί στην τσεχική πρεσβεία στις Βρυξέλλες και σήμερα εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Πολιτικές Σπουδές. Εδώ έχουμε τη Λίντα και επίσης έχουμε την Αντρέα Γκαβρίλα η οποία ε, έχει λάβει το βραβείο, έχει λάβει μια υποτροφία ε, για το Πανεπιστήμιο του Ντόν έχει εργαστεί για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Αμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κογκρέσο και έχει ουσιαστικά εργαστεί ως εθελόντρια ε, για να έχουν πρόσβαση τα θύματα εμπορίας στη δικαιοσύνη. Και Ματέι Τζούσκα, ο οποίος ε, από την Πολωνία ε, μετανάστευσε με την οικογένειά του στη Γερμανία όταν ήταν παιδί, από το 2009 έως το 2015 εργάστηκε στο Γερμανικό Μεταναστευτικό Γραφείο και έγινε πρόεδρος ε, της οργάνωσης νεολαίας της ε, ΣΕΖΗ, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων και έχει εργαστεί στην ανάπτυξη πολιτικών για τη μετανάστευση. Χωρίς χρονοτριβή, θα δώσουμε το λόγο στη Δεξίνηση με την ιδέα 1 και κατόπιν την Αντρέα για την ιδέα 2 και θα δώσω κατόπιν λόγο στους συναδέλφους. Παρακαλώ, Ματέους. Ευχαριστώ πολύ. Η πρότασή μου θα επέτρεπε σε όλες τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών της Ένωσης να λαμβάνουν αιτήσει για άσυλο ούτως ώστε να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους χρειάζονται. Θα μπορούν έτσι οι ετούντες να παίρνουν το καθεστώς του ετούντα άσυλο επίσημα χωρίς να ε, δημιουργούνται μποτιλιαρίσματα ε, από το, του, σύρους που έρχονται. Ε, μία πρεσβεία ε, μόνο λειτουργεί έτσι. Αυτό θα ήταν μεγάλη αλλαγή, γιατί θα μπορούσαμε να παρέχουμε προστασία στους ζητούντες άσυλο από την αρχή και από την άλλη οι απο, ε, θα κοινοποιούνταν στους ενδιαφερομένους ε, για να γνωρίζουν τι τύχη είχε η αίτηση. έτσι θα αποθαρρύνονταν πάρα πολύ από το επικίνδυνο ταξίδι μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στο Γερμανικό Γραφείο Μετανάστευσης είδα πολλές φορές ανθρώπους ε, που ε, έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι έγινε δεκτή η αίτηση, τους, δεν θα έκαναν το επικίνδυνο ταξίδι. Δεν θέλουμε μια κατάσταση όπου να ε, ε, ε, διακινδυνεύουν και να πεθαίνουν άνθρωποι στο ταξίδι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι μπορεί οι άνθρωποι να μπορούν να φύγουν από τη χώρα τους για να ε, τηθούν άσυλο. Οι διπλωματικές ε, αποστολές θα μπορούσαν να, να δώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και να προωθήσουν τις αιτήσει ασύλου. Έτσι θα μειωθεί η παράνομη μετανάστευση και ο ρόλος των διακινητών. Δεν είναι νέα μορφή ασύλου αυτό, αλλά έχει μακρά παράδοση στη Λατινική Αμερική και τον Καναδά. Ωραία. Και στο χρόνο πολύ ωραία, δύο λεπτά. Ελπίζω οι συνάδελφοι να τηρήσουν επίσης το χρόνο τους. Η Ανδρέα Γκαβρίλα είναι η επόμενη ομιλήτρια που θα παρουσιάσει την επόμενη ιδέα. Η Ανδρέα. Η πρότασή μου σήμερα αφορά τη δημιουργία ασφαλών ζωνών η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες ε, όπου υπάρχουν συγκρούσεις αντί για τους καταβλισμούς προσφύγων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, οι καταβλισμοί θα πρέπει να γίνουν πόλεις ασφαλείς με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι ασφαλείς πόλεις μπορούν να έρθουν σε εταιρική σχέση με Ευρωπαϊκέ πόλει, αλλά καταρχήν είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν αυτέ οι ασφαλείς ζώνες στις χώρες σύγκρουση, με το να υπάρχει στρατιωτική ασφάλεια η οποία πρέπει να γίνει σε συνεργασία με όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε και συγχρόνως τη της ε, Παγκόσμια κοινότητες. Υπάρχει μια δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Νέας Υόρκης για τους μετανάστες και πρόσφυγες που υπογράφηκε από πάνω από 190 χώρες για την ανάγκη να επανέλθει η σταθερότητα και η ασφάλεια για τους πρόσφυγες. Επίσης πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκές συγκεκριμένες δράσεις, να υπάρξουν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει καλύτερη υποδομή υγείας και εκπαίδευσης για τους πρόσφυγες και να δώσει στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε αυτές τις πόλεις τη δυνατότητα να αυτοδιακυβερνούνται και να είναι αυτάρκης. Αντί να έχουν σπίτια, να έχουν τα υλικά να φτιάξουν το σπίτι τους. Αυτοί οι οποίοι μένουν προσωρινά σε μια ασφαλή πόλη, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην υγεία και στην παιδεία, αλλά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και την προσωπικότητά τους και τη ζωή τους και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι βάσει του κράτους δικαίου και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση ή μπορούν να έχουν ένα μικρό χωράφι να καλλιεργούν. Ευχαριστώ. Έχουμε δύο ιδέες και στην ανάπτυξη, στην Επιτροπή Ανάπτυξης θα μιλήσουμε για τη Συρία σήμερα, για το πώς θα φτάσει στους δικαιούχους η ανθρωπιστική βοήθεια και φυσικά ουσιαστικά θα δούμε και πώς υλοποιείται και η δική σας ιδέα για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ε, στο πλαίσιο της μετανάστευσης βοηθά. Τι θα κάνουμε, έχουμε τρία σύνολα ιδεών, έτσι λοιπόν ε, θα το επαναλάβουμε αυτό δύο φορές. Τώρα έχουμε δύο βουλευτές ε, για ε, αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση. Η κυρία Ντεσαρμές, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με την πρώτη ιδέα που δόθηκε. Βεβαίω και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ανοίξει γραφεία έτσι ασύλου στι ε, χώρε όπου έχουμε πρόσφυγε και ιδίω για του Σύρου πρόσφυγε, στην Τουρκία, στην Ιορδανία, πιο συγκεκριμένα και στο Λίβανο. Είναι αλήθεια ότι δεν ε, είναι λογικό ότι κάποιος μπορεί να ζητήσει το δικαίωμα ασύλου μόνο αν πληρώσει τους και θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του και τη οικογένειά του για να έρθει παράνομα στην Ευρώπη, ενώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε επί τόπου. 100% συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση αυτή. Και υπενθυμίζω ότι ε, ήρθαν, έφτασαν συγγνώμη, στον Καναδά χιλιάδες άνθρωποι και ουσιαστικά η αίτηση ασύλου εξετάστηκε στις ε, γειτονικέ χώρες της Συρίας. Μπράβο λοιπόν για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Αυτό είναι κάτι που είδα όταν ήμουν στην Νότιο Τουρκία. Θα ήταν καλύτερα απευθεία ε, ουσιαστικά να συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους που να ξεκινήσουν μαζικά κύματα μετανάστευση. Ο κύριος Παντσέρη. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή αναζήτηση νέων ιδεών και ουσιαστικά φέρνει και μια ευαισθητοποίηση μεταξύ των νέων. Εγώ θα ήθελα μόνο να τονίσω τις δυσκολίες απέναντι στις ιδέες αυτές, που έχουν ιδέες αυτές. Παραδείγματο χάρη ιδέα να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές έδρες, ε, χρειάζεται να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις που σήμερα δεν φαίνονται να υπάρχουν. Καταρχήν θα πρέπει να ενισχύσουμε τις διπλωματικές έδρες που σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν ε, στο να επιτελέσουν αυτό το καθήκον. Και δεύτερον θα πρέπει να έχουμε μια διαθεσιμότητα των ευρωπαϊκών χωρών να δεχτούν τους μετανάστες. Γιατί ακούστηκε το παράδειγμα του Καναδά, είναι όμως μια χώρα, ενώ στην Ευρώπη είμαστε σε πολύ πολύ πολύπλοκη κατάσταση και όπως είδατε δεν υπάρχει αλληλεγγύη στην ανακατανομή. Και το τρίτο συστατικό είναι το εξής. Όπως ξέρετε υπάρχουν διάφορα είδη ε, τώρα έχουμε, αν έχουμε μια μεταναστευτική, μια ε, οικονομική μετανάστευση θα μπορούσαμε ε, να το αξιολογήσουμε αυτό, αλλά ουσιαστικά αυτό έρχεται σε αντίθεση με κάποιες χώρες που δεν θέλουν καθόλου τους οικονομικούς μετανάστες. Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να τους αφήσουμε σπίτι τους τους ανθρώπους αυτούς, αλλά υπάρχει και ένα άλλο είδος μετανάστευσης, οι άνθρωποι που φεύγουν από διώξεις και από εμπόλεμες περιοχές. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ε, ουσιαστικά χρονικής οργάνωσης. Δηλαδή ε, δεν είναι ότι μπορούμε να ανοίξουμε ε, ουσιαστικά τη δυνατότητα στην διπλωματικά γραφεία να πάει κάποιος ε, ε, και, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να φύγουν αμέσως. Τώρα ουσιαστικά θα μπορούσαν να διευκολυνθούν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά πρέπει να ενισχυθεί αυτή η ιδέα. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε αυτά τα συστατικά που σας ανέφερα. Ευχαριστούμε. Είναι, υπάρχουν πολλά πρακτικά θέματα για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Ας ε, κλείσουμε λοιπόν αυτό το θέμα. Η Ανδρέα θα απαντήσει στους δύο βουλευτές νομίζω ότι αφορούν περισσότερο την ιδέα του Ματέους. Εγώ θα απαντήσω για την οικονομική μετανάστευση που είναι μια μακρά αντίδραση, μακροπρόθεσμη δηλαδή και πρέπει να εστιάζει στην πρόληψη. Ευχαριστώ. Ο Ματέους. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Σάρνες που υποστήριξε την ιδέα του ΆΙ για τον κύριο Παντσέρη, σίγουρα είναι δύσκολο να αναλάβουν οι διπλωματικές αποστολές σε αυτό το καθήκον. Όπως είπα όμως στην ιδέα μου, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επιμεριστεί αυτό το καθήκον μεταξύ όλων των κρατών μελών. Ε, μία πρεσβεία στη χώρα θα μαζεύει τις αιτήσει για άσυλο και θα τις επιμερίζει. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερο προσωπικό βέβαια, είναι σίγουρο αυτό στην πρεσβεία και χρειάζονται και εκπαίδευση. Αλλά από την άλλη πλευρά αυτό που αναφέρεται ότι ένας άνθρωπος από τη, στη Συρία που έχει άμεση ανάγκη όταν ε, υποβάλλει αίτηση ασύλου στις πρεσβείες θα πρέπει άμεσα να παίρνουν κάποιον, εφοδιάζονται με ένα έγγραφο για να μπορούν να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ε, βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο μέσα από επικίνδυνα μονοπάτια. Ωραία, είναι πολύ πρακτική αυτή η ιδέα που ίσως ε, πολιτικά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί γιατί είναι δύσκολο να, ε, υπάρχει τόση συνεργασία από τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα, προγράμματα όπου έπρεπε να δεχθούμε μετανάστες ε, από καταβλισμούς που ήταν και εκεί κοντά. Ε, υπάρχει δηλαδή εμπειρία σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Η, επόμενος, ε, η επόμενη, η Λίντα Σλαπακόβα. Ευχαριστώ κυρία <clears throat> Πρόεδρε. Υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που προσπαθούν να διασχίσουν την Μεσόγειο και αυτή πρέπει να είναι και η κύρια εστίασή μας για να εμποδίσουμε τις μαζικές ροές μεταναστών. Γι' αυτό χρειάζεται ένα πλαίσιο δράση Ευρωπαϊκής Ένωση Μεσογείου για να αντιμετωπίσει τι ανάγκε των ε, ανθρώπων αυτών, των νέων ανθρώπων στι χώρε αυτέ, κυρίως με περισσότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγεία, κυρίως το να δώσουμε ευκαιρίες σε αυτούς, γιατί η έλλειψη ευκαιριών από του κύριου λόγου τη μετανάστευση, αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, με μακροχρόνια προοπτική θα αναγκαστούν και πάλι να φύγουν αυτοί από τις χώρες, σας, από τις χώρες τους για να βρουν κάποιες ευκαιρίες. Δεύτερον, μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ οργανώσεων των νέων και κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη και αλλού για να αντιμετωπίσουμε τον βίο εξτρεμισμό και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά τους. Εγώ μπορώ να πω ότι ο βίος εξτρεμισμός και η ριζοσπαστικοποίηση, η άκρα ριζοσπαστικοποίηση οδηγεί σε ε, ακραίες καταστάσεις και ανασφάλεια. Γι' αυτό όλη η διεθνή κοινότητα πρέπει να αντιμετωπίσει τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση και να σταματήσει τη βία με προγράμματα όπως αυτά που υποστηρίζουν την κοινωνία των πολιτών και αυτό μπορεί να εξαχθεί και στην νότια οχθή της Μεσογείου. Επίσης να δημιουργήσουμε από στελεσματικά προγράμματα επανενσωμάτωσης για τους μετανάστες που γυρίζουν στις χώρες τους, ώστε να γίνουν πιο περιεκτικές τοπικές κοινωνίες και να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο στο οποίο οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Αντρέα Καβρίλα θα μας, φέρει, θα μας δώσει τη δεύτερη ιδέα στο θέμα αυτό. Βασιζόμενοι στην αρχή ότι αν δώσετε, μάθετε κάποιον να ψαρεύει θα ψαρεύει όλη τη ζωή και δεν χρειάζεται να του δίνετε ψάρια, εγώ θεωρώ ότι οι επιτροπές ΔΕΒΕ και ΑΦΕΤ θα πρέπει να φτιάξουν ένα σώμα νέων. Ένα σώμα για την ειρήνη από τους νέους. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους να αναπτύξουν στις τοπικές τους κοινότητες τις δικές τους ικανότητες και να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή ατζέντα για την μετανάστευση αυτοί οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν μπορούν να πάνε στις αναπτυσσόμενες χώρες και να δώσουν στον τοπικό πληθυσμό τις δεξιότητές τους για τη γεωργία, για την πράσινη ενέργεια κτλ. Γνωρίζετε ότι μπορεί να φτιάξει κανείς ένα ανεμόμυλο από ένα κατεστραμμένο ποδήλατο, αλλά εγώ το είδα από τα μέσα ενημέρωσης όταν κάποιος στο Μαλάουε έχει φτιάξει ηλεκτρικούς ε, ανεμόμυλους, μάλλον ανεμόμυλους που παράγουν ηλεκτρισμό από απλά υλικά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει αυτό σε τοπικές κοινότητες για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι συγκρούσεων και να υπάρχουν κέντρα για τους νέους. Θα πρέπει να δοθεί σε αυτούς τους νέους ένα βασικό εισόδημα και χρήματα για την εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο και αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να υποστηριχθεί. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι αντικείμενα αναφορών και να γίνουν ορατά για να είναι και ένα παράδειγμα για τους άλλους. Και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τους νέους να έχουν μια ζωή η οποία θα έχει κάποιο νόημα και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί ο ριζοσπαστισμός και ο εξτρεμισμός μπορεί να του οδηγήσει σε, στο θάνατο και μόνο. Ευχαριστώ συνάδελφε έχετε κάποιες ε, απαντήσεις σε αυτές τις ιδέες. Εδώ ακούσαμε το, την υποστήριξη των νέων να συνεργαστούν μαζί τους για να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα. Ξέρουμε ότι στην Αφρική η δημογραφική η ανάπτυξη είναι τεράστια πρόκληση σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασία. Και χθε ακούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση στην Επιτροπή Ανάπτυξη για τα μικρά χωριά, πώ τα αφρικανικά χωριά αναπτύσσουν οι άνθρωποι λύσει εκτό δικτύου για την παραγωγή ενέργεια. Και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και πέφτει το σκοτάδι στι 6 το βράδυ. Έτσι λοιπόν και το θέμα τη μεταφορά τεχνολογική γνώση είναι στην υπηρεσία διάταξη. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να αντιδράσουν σε αυτές τις δύο ιδέες, κάποιοι βουλευτές. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ε, ιδέες σας ε, και που ήρθατε εδώ να μας τις παρουσιάσετε. Να προσθέσω κάτι. Έφτασα καθυστερημένη για τη μουσέλη συνεδρίαση. Ίσως να καλύψατε ήδη αυτό το θέμα όμως. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο αγωνιζόμαστε και για πολλά χρόνια, τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, ζητάμε μία λύση ε, έτσι ώστε να υπάρχουν κοινέ προσπάθειε μεταξύ των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πριν δύο εβδομάδε ήμουν στη Νέα Υόρκη, είχαμε την πρώτη σύνοδο σε επίπεδο ΙΕ για τη μεγάλη μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών. Και φυσικά εκεί συζητήσαμε για μια παγκόσμια προσπάθεια που χρειάζεται να γίνει, γιατί η μετανάστευση και η υποδοχή των προσφύγων είναι παγκοσμία πρόκληση και χρειάζονται φυσικά παγκοσμίες λύσεις, αλλά πόσο αξιόπιστοι μπορούμε να είμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, ε, εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν μπορούμε να έχουμε κοινέ λύσει που χρειαζόμαστε απελπισμένα, γιατί σήμερα έχουμε 6 από τα 28 κράτη-μέλη που μόνα του προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το 80% των αιτήσεων ασύλων που κατατίθεται στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι βιώσιμο για κανέναν. Αλλά όπω σε κάθε προσπάθεια, αν ε, μπορεί να, να την επιμερίσουμε στους 28 θα είναι βιώσιμη για όλους. Αυτό υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι πολύ σημαντικό. Εμείς ως βουλευτές επιστρέφουμε στις πατρίδες μας σχεδόν κάθε εβδομάδα και προσπαθούμε να εξηγήσουμε και προσπαθούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τους συμπολίτε μας στις πατρίδες μας. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να κατανοήσει κανείς τις διάφορες ευθύνες μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις διάφορες αρμοδιότητες. Όμως πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την επιμερισμένη προσπάθεια, γι' αυτό διαφορετικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οι αναγόμες. Και εγώ λυπάμαι που δεν μπόρεσα να ακούσω όσο υπόθηκαν, γιατί ήρθα καθυστερημένη από μια άλλη συνεδρίαση, αλλά άκουσα το τέλος των παρεμβάσεων και πραγματικά ε, ήταν πολύ στοχευμένα όσα υπόθηκαν. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους να είναι ενεργοί και να προωθούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό με οδηγεί στον να το εξής την ανάγκη ε, πάνδρωσης. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις μας ε, να επενδύσουν στρατηγικά σε προγράμματα προκειμένου να καταπολεμήσουν τη διάδοση των εξτρεμιστικών ιδεολογιών που οδηγούν στη βία. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει αρκετή δουλειά της κυβερνήσης μας στον τομέα αυτό. Εμείς σε αυτό το κοινοβούλιο, εδώ και πολύ καιρό, πριν ένα έτος, αναφέραμε το θέμα της πρόληψης. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγες οι επενδύσεις και οι επενδύσεις αυτές δεν θα λειτουργήσουν αν δεν εμπλακούν και οι νέοι, οι ενώσεις των νέων σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να μπορούν να είναι πραγματικοί πρωταγωνιστές για να καταπολεμήσουν αυτή την ιδεολογία των τρομοκρατικών ομάδων. που δυστυχώς οδηγεί σε περισσότερη βία. Φυσικά πρέπει να έχουμε και πολιτικές πραγματικά να δίνουν αρμοδιότητες στους νέους και θα πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικές ευκαιρίες, δουλειές, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι θα κάνουμε καλή δουλειά και θα έχουμε καλά αποτελέσματα το τομέα της πρόληψης αν ταυτόχρονα δεν προσφέρουμε βασικές ευκαιρίες στους νέους, δηλαδή δημιουργία θέσεων εργασία κτλ. Και ουσιαστικά πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτές τις ηλίθιες πολιτικές λιτότητας που υποσκάπτουν και τη δική μας ασφάλεια και θα πρέπει να έχουμε κοινωνική ολοκλήρωση. Επίσης, συμφωνώ με όσο είπε η Έλλη για το θέμα των προσφύγων όπως οι κυβερνήσεις μας διαχειρίζονται την εισρωή προσφύγων και μεταναστών. Δεν θα σταματήσει φυσικά αυτό με φράκτες πολέμους. Θα έρχονται και όλο και περισσότεροι θα έρχονται και ουσιαστικά η Ευρώπη θα πρέπει να όσο μάλλον δεν παρεμβαίνει για την επίλυση της ε, σύραξης τόσο περισσότεροι θα έρχονται έχουμε ε, θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση που δεν θα συνεχίσει να δίνει δουλειά στους δουλεμπορούς. Ε, και ο Αντώνιο Γκουτιέρες είπε, ξέρουν ε, οι δουλεμποροί πώς να διαχειριστούν την ροή των προσφύγων. Εμείς είμαστε αυτοί που δεν το κάνουμε αυτό, γιατί κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά δίνουμε και βοηθάμε τους ανθρώπους αυτούς ε, να έχουν δουλειά. Ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε ε, ουσιαστικά τη δουλειά των δουλεμπόρων είναι να ανοίξουμε νόμιμες και ασφαλείς οδούς για τους ανθρώπους να μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι είτε ως πρόσφυγες και να ζητήσουν προστασία είτε ως μετανάστες. Όσο αρνούνται οι κυβερνήσεις να το κάνουμε αυτό, τότε θα δίνουμε δουλειά στους διακινητές και πρέπει οι νέοι να υψώσουν τη φωνή τους και να μιλήσουν γι' αυτό. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Να ακούσουμε τις επόμενες δύο ιδέες και μετά να σχολιάσετε στο τέλος, αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Πάμε λοιπόν στις επόμενες δύο ιδέες. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει να σχολιάσει ε, και να αντιδράσει αυτά που ακούσαμε για τους νέους και το Ευρωπαϊκό Θελοντικό Πρόγραμμα. δεν ξέρω αν συζητήσατε στο Στρασβούργο όταν έγινε η εκδήλωση. Ε, η Λίντα θα παρουσιάσει τώρα μια άλλη ιδέα. Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρεται στις τελευταίες ε, παρεμβάσεις για τη διακίνηση ανθρώπων και την εφαρμογή του νόμου. Η τελευταία έκθεση Europol έδειξε ότι στο επίκεντρο του προβλήματος ε, ε, είναι ένα δίκτυο που το αξιοποιεί το 90% των παράνομων μεταναστών. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν να βρεθούν νόμιμες, νόμιμοι διάβλοι. Μπορούν να γίνουν περισσότερα για την εφαρμογή του νόμου και για την προστασία των συνόρων έτσι. Ε, θα καταπολεμηθεί και το οργανωμένο έγκλημα. Η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης και τρίτων χωρών είναι σημαντική. Υπάρχουν πλατφόρμες συνεργασίας μεταξύ κρατών και ε, οργανισμός Europol, Eurojust, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα στις τρίτες χώρες και γι' αυτό χρειάζονται πιο πολλά πράγματα για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τρίτων Χωρών και Κρατών Μελών για την καταπολέμηση αποτελεσματικότερα του οργανωμένου εγκλήματο. Ε, τελευταία υπάρχει, έχει δημιουργηθεί το κέντρο ε, κατά της διακίνησης ε, ανθρώπων. Είναι σημαντικό να γίνει και αλλού και θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη Μεσόγειο που εκεί υπάρχει μια πολυμερής ε, πλατφόρμα συνεργασίας πολλών χωρών. Ε, αυτό είχε αναφερθεί και στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας στα Βαλκάνια. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα δημιουργεί ένα αφήγημα ε, χωρίς να θεωρεί τους μετανάστες υπέτειους για κρούσματα βίας ε, υπάρχουν τέτοια αφηγήματα παντού. Ο στιγματισμός ως εγκληματιών των μεταναστών ε, έπαιξε πολύ κακό ρόλο. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφές το αφήγημα. Δεν είναι οι, οι ε, παράνομοι οι μετανάστες, ε, δεν είναι οι εγκληματίες εκείνοι, αλλά εκείνοι που τους εκμεταλλεύονται από το οργανωμένο έγκλημα. Ο η δεύτερη μου πρόταση είναι να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων όπου θα υποβάλουν το βιογραφικό τους οι μετανάστες για να διαπιστωθεί αν έχουν δεξιότητες που χρειάζονται στις χώρες ε, που θέλουν να μεταναστεύσουν θα υποβάλλεται αίτηση στο κράτος μέλος, το κράτος μέλος θα ε, παληθεύει την ε, αίτηση, θα την επιβεβαιώνει και θα ενημερώνει αν υπάρχει ενδεχόμενο απασχόληση ε, από για το μετανάστη ανάλογα με γλώσσες, ε, ε δεξιότητες κλπ. Είναι πιο σημαντικό να, βλέπω, ε, να, να ακολουθεί μια τέτοια διαδικασία και για το κράτος μέλος και για το μετανάστη. Θα πρέπει να ε, λαμβάνει την υπόψη και η βούληση του μετανάστη αλλά και οι ικανότητες ένταξης από τη χώρα μέλος. Έτσι θα είναι πολύ πιο διαφανής η διαδικασία εισόδου. Ο συνδικαλιστής ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μπει κανείς στη σημερινή αγορά εργασίας. Ακόμα και οι μεδαποί δυσκολεύονται όταν πρόκειται για μετανάστες. Τα προβλήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα αφού πρέπει να ξεπεράσουν γλωσσικούς φραγμούς, ε, δεν ξέρουν αν θα αναγνωριστούν οι δεξιότητες ε, και αυτό ε, δημιουργεί έλλειψη αυτοπεποίθησης. Οι χώρε υποδοχή θα πρέπει να δίνουν στου μετανάστε λοιπόν και καλή επιμόρφωση, ε, κατάρτιση για να μπουν στην αγορά εργασία. Και έτσι περνώ σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τη ένταξη Ενσωμάτωση ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας. Ε, θα πρέπει να αναγνωριστούν ε, τα προσόντα που έχουν ήδη. Πολλές φορές είναι υψηλή εξειδίκευση και δεν αξιοποιούνται γιατί δεν αναγνωρίζονται προσόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ε, εκπαιδευτεί αλλού. Χρειάζεται ένα σύστημα ισοδυναμίας των διπλωμάτων, συστήματα πιστοποίηση που να αναγνωρίζονται από τη χώρα υποδοχής. Για να επιτύχει ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στον δημόσιο τομέα, στις δημόσιες υπηρεσίες δηλαδή. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να απαντήσει, να αντιδράσει σε αυτές τις τελευταίες δύο ιδέες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Χιμένεθ. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση γιατί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως είναι το θέμα της μετανάστευσης, κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τους απλούς ανθρώπους και τους νέους. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συνεδρία. Είναι πολύ καλό το ότι γίνεται και με την παρουσία και των δύο επιτροπών της ΑΦΕΤ και της ΔΕΒΕ. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο εδώ πέρα να ενισχύσουμε είναι η αξιοπιστία της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό θέμα γιατί εδώ παίζεται όλο το παιχνίδι γιατί οι πολίτες περιμένουν απαντήσεις και για την ασφάλεια και για την τρομοκρατία και την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και της κρίσης των προσφύγων που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή στα μάτια των νέων διακυβεύει το κατά πόσο θα θεωρήσουν ότι αξίζει τον κόπο να αγωνιστούν για την Ευρώπη. Η Υπηρεσία Εξωτερικών Εξωτερικής Δράσης έχει τονίσει την ε, ανάγκη αλληλεγγύης και προς τις χώρες που βρίσκονται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιο είναι το μήνυμα που θα δώσουμε στους νέους, κατά πόσο είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε μεταξύ μας σε ένα τόσο κέριο αλλά και δύσκολο θέμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε <clears throat> το θέμα της ε, πηγής αυτών των ροών. Αυτό δεν μπορεί να επιληθεί από την Ευρώπη την ίδια η Ευρώπη δεν μπορεί να τα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στις χώρες προέλευσης, στη ρίζα του προβλήματος. Και έχουμε το πρόβλημα των ε, διακινητών που χρησιμοποιούν τους ανθρώπους σαν να είναι εμπορεύματα και προσπορίζονται εκατομμύρια και εκατομμύρια. Πέραν των εκθέσεων που έχουμε κάνει και όλων αυτών που έχουμε τονίσει. Δεν έχουμε ασκήσει πραγματική πίεση για να αντιμετωπίσουμε <clears throat> το πραγματικό πρόβλημα που είναι ότι ασκείται αυτή τη στιγμή ένα παράνομο εμπόριο ανθρώπων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να σταθούμε στο θέμα της διακίνησης ατόμων και επίσης να αντιμετωπίσουμε και τη ρίζα του προβλήματος γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο μπορούμε να ζητάμε, να προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, να ζητήσουμε το φεγγάρι και τα άστρα δεν θα πετύχουμε τίποτα. Χρειάζεται αλληλεγγύη και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή θέση και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν, είπα, δεν είδα κάποιον άλλο που θέλει να ε, πει κάτι. Ίσως κάποια τελικά σχόλια για, τα δύο αυτά, για τις δύο αυτές ιδέες. Η Λίντα πρώτα. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το αφήγημα το οποίο διαδίδει προς τους πολίτες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λένε ότι οι συμφωνίες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται για το συμφέρον της. <clears throat> Αυτό όμως δημιουργεί μια αρνητική κατάσταση που οδηγεί τους νέους οι οποίοι περιμένουν μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να απογοητεύονται μπορεί η κατάσταση να βελτιωθεί στο μέλλον. Αλλά αν δίνεται σαν προτεραιότητα αυτές τις ε, συμφωνίες, αυτό σημαίνει ότι υποχωρεί σε σχέση με τις αξίες της Ευρωπαϊκή Ένωση και ασχολείται μονάχα με το θέμα της ασφάλειας. Αν δεν υπάρξει καλύτερη ασφάλεια και καλύτερη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη σχέση μας με τις χώρες της ε, νότιας όχθης της Μεσογείου και της Αφρικής. Όλα αυτά λοιπόν είναι η ουσία του προβλήματος. Είναι θέμα πολιτικής θέλησης για μένα. Και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια συνεκτική στάση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αντρέα. Θα ήθελα να απαντήσω στα προηγούμενα σχόλια Πράγματι, υπάρχει πρόβλημα με το ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπαθίες μας. Κατά κάποιο τρόπο είναι λογικό να υπάρχουν αποκλίνωσες ε, απόψη, όμως ε, το σύνθημά μας ε, είναι ενωμένοι στην ποικιλομορφία. Πώς φτάνουμε λοιπόν σε αυτή την ενότητα. Νομίζω ότι μία από τις ε, λύσεις ε, και πάλι έγκυται στους νέους, γιατί ουσιαστικά συναντιούνται πιο εύκολα και δέχονται πιο εύκολα τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσετε να επενδύετε σε προγράμματα για την νεολαία, γιατί όταν εμπλέκετε τους νέους, τους δίνετε και νόημα. Παραδείγματο χάρη, η σημερινή εμπειρία είναι πολύ σημαντική για μα, προκειμένου να δούμε ότι μα ακούνε και μάλιστα είμαστε ακόμη και πιο ενθουσιώδει όταν βλέπουμε ότι θα γίνουν πραγματικότητα κάποιε από αυτέ τι ιδέε. Ας μην ξεχνάμε ότι ένας οίκος χωρίς ενότητα είναι οίκος χωρίς δύναμη, χωρίς εξουσία. Έτσι λοιπόν, ας δώσουμε δύναμη σε αυτόν τον οίκο. Ο Ματέους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που συμφωνείτε. Χαιρόμαστε που ακούμε ότι σας αρέσουν οι ιδέες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ακόμη πιο ισχυρή και να δείξει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεργαστούν προκειμένου να επιλύσουν το μεταναστευτικό πρόβλημα. Καθώς εμείς οι τρεις εκπροσωπούμε τη μεγαλύτερη εκδήλωση της νεολαίας και εκπροσωπούμε την νεολαία της Ευρώπης, νομίζω ότι σας δείξαμε ότι θέλουμε μια Ευρώπη που να στέκεται ενωμένη, να είναι ελεγγύα και θέλουμε οι νέοι να έχουν φωνή και φυσικά να ακούγεται η φωνή τους. Σας ευχαριστώ. Να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αντιδράσει. Το πολύ δύο λεπτά παρακαλώ. Μαρία Τεπαόλης, παρακαλώ. Δεν ξέρω που κάθεστε. Εκεί κάτω. Ευχαριστώ Μαρία. Ε, μετά Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη η ΔΕΦΚΟ αντιμετωπίζει τις ε, αιτίες της μετανάστευσης. Μπορώ να αναφέρω κάποια παραδείγματα εφαρμόζουμε δράσεις για να δώσουμε ε, εξουσίες, αρμοδιότητες στην νεολαία σε κάποιες χώρες, χώρες για να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εφαρμόζουμε προγράμματα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και αναλύουμε τις δυνατότητες να βελτιώσουμε την αγορά εργασίας και να αποφύγουμε τις αναντιστοιχίες μεταξύ της ε, εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Επίσης, ε, θα έχουμε να αναγνωρίζονται τα προσόντα στις χώρες εταίρους, προκειμένου να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα μεταξύ των χωρών. Και φυσικά σε ό,τι αφορά τις αιτίε, ε, δεν ε, πρέπει να εστιαστούμε μόνο αυτό. Ε, πρέπει ουσιαστικά να δούμε ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι από την παιδική τους ηλικία. Τα σημερινά παιδιά θα γίνουν η επόμενη γενιά μεταναστών. Και βλέπουμε πολλά παιδιά μετανάστες να έρχονται στην Ευρώπη ασυνόδευτα. Και είναι σε πάρα πολύ ευάλωτη κατάσταση. Επομένως, έχουμε μία σειρά δράσεων στην Κομισιόν που στοχεύουν στο να διασφαλίσουν τη συνεκτικότητα, αλλά κάνουμε και μία αποτίμηση άλλων πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης συνεργαζόμαστε με το ΕΚΟ, το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοηθείας, για να προσφέρουμε εκπαίδευση, υπηρεσίε υγεία και όλες τις βασικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητε στους πρόσφυγες. Αυτά είναι μόνο κάποια παραδείγματα. Αν χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθεία σε εμά. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους μας σήμερα. Βλέπετε ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να βρουν λύσεις για το μεταναστευτικό, αλλά πολλές φορές μπλοκάρουν τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν πολλά δύσκολα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, η κοινή γνώμη και ε, εδώ βέβαια καλό είναι που μας ενημερώσατε, αλλά καλό είναι να διαμορφώνεται και συνένεση μέσα από τη δική σας προσπάθεια και στις χώρες μέλη. Ε, θα πρέπει να δοθεί μάχη σε κάθε επίπεδο για μια πιο συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Να ευχαριστήσω με πάρα πολύ λοιπόν τους προσκεκλημένους μας που ήρθαν με τις ιδέες τους εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι καλή ιδέα ότι ακούσαμε περισσότεροι ε, από διάφορες επιτροπές τις προτάσεις σας. Ελπίζω ότι ε, στην επόμενη συζήτηση θα ε, ληφθούν υπόψη και άλλες ιδέες για τη μετανάστευση. Προχωράμε τώρα στο σημείο 13, κοινή έκθεση μεταξύ της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το άρθρο 35 είναι μια ε, έκθεση σχετικά ε, με την ε, ευρωπαϊκή εξωτερική δράση το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα μετανάστευσης και ε, μεταναστών και προσφύγων. Είναι μια διάσταση της εξωτερικής πολιτικής. Οι δύο επιτροπές μας ε, συμμετέχουν πολύ, ε, υπάρχουν τα, έχουν ασχοληθεί με τα σύμφωνα μετανάστευσης. η συζήτηση την περασμένη εβδομάδα για το δρόμο και το τι θα γίνει μπροστά. Ε, διάφορα θέματα μας έχουν απασχολήσει στα πλαίσια της πολιτικής εξωτερικών υποθέσεων και ε, ε, ανάπτυξης. Η αναπτυξιακή χρηματοδότηση κινητοποιήθηκε για να λυθούν κάποια προβλήματα σχετικά με το μεταναστευτικό. Είναι καλό που υπάρχει κοινή έκθεση. Έχουμε την Ελένα Βαλενσιάνο και τον Ογκουστίν Δίας Δεμέρα, συνεισηγητές που είναι και οι δύο εδώ. Ε, υπάρχει η έκθεση στο φάκελό σας με ορισμένες ιδέες. Δεν ξέρω με ποια σειρά θα τα τους πάρουμε. Ίσως πρώτα να ακούσουμε την Ελένα Βαλενσιάνο και μετά τον Ογκοστίν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακολουθώντας το οδηγό των, ε, αυτών που είπατε προηγουμένως, προφανώς έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλία η οποία δεν θα αλλάξει αφ' αυτή στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά της μετανάστευσης. Είναι γεγονός ότι το εργαλείο της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει όλο και περισσότερο υπόψη τα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η Επιτροπή με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να ακούσει κάποιες από τις απόψεις της Επιτροπής Ανάπτυξης που εξάλλου νομίζω ότι τις συμμεριζόνται πάρα πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεγάλα στρώματα του πληθυσμού συμφωνούν με αυτές τις ιδέες. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το θετικό πνεύμα που έδειξε ο κύριος Δίας μέρα για μια έκθεση η οποία δεν ήταν εύκολη έκθεση γιατί όταν δουλεύουν δύο επιτροπές πάνω στο ίδιο θέμα αυξάνεται η πολυπλοκότητα της προετοιμασίας μιας έκθεσης αλλά εμπλουτίζεται και η συζήτηση. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα αλλά πρέπει να πω ότι ήταν πολύ καλή συνεργασία μας με τον κύριο Στεμέρα και μπορέσαμε να επιτύχουμε μια πολύ σημαντική συνένεση και βάση για να δώσουμε τα μηνύματα που πρέπει να δώσουμε. Όπως γνωρίζετε όλοι, το περιθώριο για μια έκθεση πρωτοβουλία είναι περιορισμένο, γι' αυτό κάναμε και μια παράλληλη έκθεση που απαρτίζεται από ένα σύνολο τροπολογιών που για λόγους χώρου περιορισμένη έκταση δεν μπορούν να περιληφθούν στην έκθεση, αλλά και που υποστηρίχθηκαν και από τους δύο εισηγητέ. Πέρα λοιπόν αυτών των τεχνικών ζητημάτων, θα ήθελα να σταθώ σε δυο τρει ιδέε, οι οποίες είναι αυτέ που περιλαμβάνονται στην έκθεσή μας. Και είναι το πνεύμα με το, από το οποίο εμφορείται η έκθεσή μα. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί αυτή τη στιγμή προς μια αντίληψη του φαινομένου μετανάστευσης ή αν θέλετε της κινητικότητας των ανθρώπων που είναι πολλές φορές αντιφατική προσέγγιση. Πολλές φορές η αν της κινητικοτητας των ανθρωπων που ειναι πολλες φορες αντιφατικη προσεγγιση πολλες φορες η προσεγγιση μας είναι καθαρά αμυντική, να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές, να κλείσουμε τα σύνορά μας στο βαθμό του δυνατού, να εμποδίσουμε την είσοδο αυτών των ανθρώπων, ενώ συγχρόνως και παράλληλα υπάρχει μια ηθική και πολιτική ανησυχία πολλών ανθρώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά και της κοινή γνώμης που λέει ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο δεκτικοί να υποδεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους, να δώσουμε την δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν στην Ευρώπη γιατί οι μετακινήσεις των λαών <clears throat> έχουν δημιουργήσει και τον πολιτισμό στον οποίο ζούμε. Θα πρέπει λοιπόν να μην εμποδίσουμε αυτές τις ροές των ανθρώπων αυτών. Κάποιες από αυτές τις κινήσεις έχουν μια τυποποίηση και μια ε, νομική βάση, αν θέλετε, στο διεθνές δίκαιο, ακόμα και αν δεν τηρούμε εμείς στο διεθνές δίκαιο. Κάθε κατηγορία ανθρώπων, λοιπόν, που εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες πρέπει να τύχει κάποιε προστασίε. Κυρίω πρόκειται για ανθρώπου που πρέπει να φύγουν από τη χώρα του και να βρουν μια καλύτερη ζωή, κάποια ψήγματα αξιοπρέπεια στη ζωή του. Και τώρα σε αυτή την αντίφαση μεταξύ του, της, αντιμετώπισης, της αντιμετώπισης των ροών των ανθρώπων αυτών που μετακινούνται και συγχρόνως να σεβαστούμε τις αξίες που απετέλεσαν τη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρισκόμαστε σε αυτή την κατά κάποιο τρόπο διχασμένη προσέγγιση. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε υπερβολικά προς την κατεύθυνση της αμυντικής διαχείρισης των ροών, ενώ θα πρέπει να δείξουμε κάποια ενσυναίσθηση, κάποια ανθρωπιστική αντιμετώπιση, κάτι το οποίο σε πολιτικό επίπεδο είναι απαραίτητο αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις αρχές από τις οποίες έχει εμπνευστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται προσπάθειες σε πολλά επίπεδα με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι στις πηγές των ε, μετακινήσεων αυτών, στις χώρες από όπου φεύγουν ε, οι αυτοί οι άνθρωποι, θα μπορέσει να υπάρξει κάποια λύση, κάποιο σύστημα που θα τους ε, δώσει λιγότερο κίνητρο να φύγουν από τη χώρα τους. Αλλά οι συμφωνίες οι οποίες γίνονται με τρίτες χώρες μας οδηγούν σε πολλές αμφιβολίες και ανησυχίες. Και σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν γνωρίζει πολύ καλά τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτές οι συμφωνίες. Οι συμφωνίες λοιπόν αυτές είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από την θέση που μπορεί να έχει το Κοινοβούλιο και από τον έλεγχο ο οποίος κανονικά ανήκει, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν κάποια κονδύλια αναπτυξιακά που δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για αυτό το λόγο για την συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση είναι δύσκολη γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε τα πράγματα να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο που οι αποφάσει οι οποίε ελέγχθηκαν στη συνέχεια δεν ήταν οι καλύτερε δυνατέ αποφάσει και αυτό γίνεται όταν αφήνουμε ένα τρενάρι, ένα πρόβλημα, καταλήγουμε σε λύσει οι οποίε δεν είναι οι καλύτερε, είναι χειρότερε από ό,τι αν είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην αρχή του. Γι' αυτό τονίζω ότι μα απασχολούν πολύ ορισμένα από τα μέτρα τα οποία προτείνονται και πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δείξει μεγάλη προσοχή σε όλα αυτά που γίνονται. Υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες που δεν ε, μας εξηγούν πώς θα πρέπει να γίνονται οι συμφωνίες αυτές παραγωγή για την περίπτωση του Αφγανιστάν, η συμφωνία επανιστοχής για το Αφγανιστάν. Μιλάμε για 80.000 άτομα τα οποία θα επαναποσταλούν στο Αφγανιστάν. Θα θέλαμε να ξέρουμε πώς θα τους επανενσωματώσει το Αφγανιστάν. Ξέρουμε ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν καμία δυνατότητα να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Έχουν ανάγκη κάποιας βοήθειας από τις κυβερνήσεις των χωρών μας που έχουν συνάψει αυτές τις συμφωνίες. Φυσικά δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε μόνο μια κριτική κενή νοήματος. Θα πρέπει να υποβάλουμε και θετικές προτάσεις, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να θέσουμε στο προσκήνιο τις αρχές και τις αξίες μας, οι οποίες θα πρέπει να διέπουν τη δράση μας σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές. Και οι αρχές αυτές βρίσκονται μέσα στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό το οποίο εδώ και πολύ καιρό από πολλές πλευρές το τονίζει η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν ένα αφήγημα το οποίο είναι τελείως αρνητικό σε σχέση με το, με το φαινόμενο της μετανάστευσης και έχουν δημιουργηθεί προστοκίες με τα ταμεία αυτά τα οποία έχουν προταθεί να δημιουργηθούν και που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν στην πράξη. Εγώ υποστηρίζω λοιπόν και τις προσπάθειες της Κομισιόν και τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης για να δημιουργηθεί μια πραγματική εξωτερική πολιτική για το θέμα της μετανάστευσης. Είναι κάτι το οποίο μας λείπει. Χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική μετανάστευση, η οποία όμως έχει να έχει και στατηγικό χαρακτήρα να <clears throat> βασίζεται σε αρχές και να εδράζεται στην κοινή ευθύνη και την αλληλεγγύη. Υπάρχουν πολλά περισσότερα ερωτήματα για τα οποία μπορούμε, όπου μπορούμε να σταθούμε, να τα αντιμετωπίσουμε τις ε, βασικές αιτίες μετανάστευσης, να έχουμε νόμιμη μετανάστευση για να αντιμετωπίσουμε την παράνομη διακίνηση, μια κοινή θέση με τις ε, τρίτες χώρες από όπου προέρχονται οι μετανάστες για να μην επιβάλλουμε στη τη θέλησή μας αλλά να είναι μια κοινή συμφωνία να λάβουμε υπόψη και τον ρόλο των γυναικών γιατί οι γυναίκες όχι μόνο υποφέρουν περισσότερο αλλά μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο για να μειωθεί η μεταναστευτική ροή και νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να ενισχυθούν με τις απόψεις που θα μας δώσουν και οι συνάδελφοι και με τη βελτίωση με τι τροπολογίε του κειμένου μα. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση από κάθε άποψη, γιατί μονάχα με μια εξωτερική δράση η οποία θα είναι αποτελεσματική, θα είναι στεναρή, θα είναι ισχυρή και εδρεωμένη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με αξιοπρεπή τρόπο την κινητικότητα των ανθρώπων στον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριος Δίας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Λίντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Ελένα. Και εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ άνετα στα πλαίσια της συνεργασίας μας και εκτιμώ τις ιδέες της. Στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και προσπαθώ να τις εναρμονίσω με το πλαίσιο των δικών μου αρμοδιοτήτων. Έτσι λοιπόν, εδώ αναφέρομαι στην πολιτική ανάπτυξη. Η εξωτερική δράση και ανάπτυξη έχουν μια άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Και εμείς προσπαθήσαμε να τονίσουμε αυτή τη σχέση μέσω μιας διπλής έκθεσης η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει η μία με τον κανονισμό και είναι πιο συνοπτική και η άλλη έκθεση είναι πιο εκτεταμένη σε σχέση με την προοπτική των πρωτοβουλίων μας, χωρίς νομοθετικό περιεχόμενο. Εκεί όμως παρουσιάζεται μια ιδεολογική φιλοσοφική θέση επί του θέματος. Η συνάδελφος αναφέρθηκε ήδη εκτεταμένα στο θέμα αυτό, το εξήγησε με σαφήνεια. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες πιο συγκεκριμένες πτυχές της έκθεσης. Όμως, πρέπει να πω καταρχήν ότι χθε είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον Πέρο Λουκ, με τον Ρίκε Γκερέρο, με τον κύριο Πάβο και με τη Χέντι Χαουτάλα τις ε, πρώτες ιδέες μας. Ε, ήταν ιδιαίτερα πλούσια η συνάντηση αυτή, γιατί οι συνάδελφοι παρουσίασαν μία σειρά ανησυχιών που έχουν και που μπορούν να εμπλωτίσουν τη δουλειά που κάνουμε εγώ και η Ελένα. Γι' αυτό σας ε, καλώ μέχρι τις 18 εντός της προθεσμίας να παρουσιάσετε και τις δικές σας συνεισφορές. Εμείς έχουμε διαιρέσει την έκθεσή μας σε τέσσερα μέρη. Το ένα μέρος έχει να κάνει με την παγκόσμια δράση και τις αρχές ε, της Ένωσης για να απαντήσει στις προκλήσεις της κινητικότητας. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με τη διεθνή μετανάστευση, που θα είναι διεθνή μετανάστευση από καλύτερη διαχείριση και στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας ευθύνης. Το τρίτο τμήμα έχει να κάνει με την εξωτερική δράση της Ένωσης συγκεκριμένα και τις συμφωνίες συνεργασίας και σύνδεσης με τρίτες χώρες και το τέταρτο μέρος αφορά τα κατάλληλα μέσα για τις δράσεις που προτείνουμε. Εμείς ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ροές είναι παγκόσμια ευθύνη και επομένως απαιτούν και μια παγκόσμια λύση και μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων κρατών. Ήδη αυτό τονίστηκε στη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου των, ε, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου συζητήθηκαν ακριβώς οι μεγάλες ροές των προσφύγων και μεταναστών ε, στις, ε, και στην ε, Σύνοδο Κορφής που οργανώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμετείχαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάθε απάντηση σε αυτές τις μεταναστευτικές ροές θα πρέπει να γίνει υπό την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων. Αυτό διέπει όλες μας τις πολιτικές γιατί η χάρτα είναι πρωτογενές δίκαιο και ό,τι κάνουμε στο νομοθετικό πεδίο ή όχι θα πρέπει να σέβεται το πρωτογενές δίκαιο που υπάρχει στη χάρτα. Τονίζουμε ως πολύ σημαντικό το ρόλο των γυναικών σε σχέση με τις αναγκαστικές μετακινήσεις και υπενθυμίζουμε ότι τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι είναι σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες τους έναντι των ε, επαναλαμβανόμενων καταχρήσεων. Επίσης, επενθυμίζουμε ότι μια καλή διαχείριση στο μεταναστευτικό συνεισφέρει σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Όπως Ελένα και επαναλαμβάνω και εγώ, θα πρέπει να αλλάξουμε την σημερινή αφήγηση, η οποία είναι πάρα πολύ αρνητική, και να διευκολύνουμε μία κατανόηση του φαινομένου πολύ πιο θετική. Για να το πετύχουμε είναι απαραίτητη να υπάρχει μία κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική με νόμιμες διόδους για τη μετανάστευση. Δεν θέλω να σας κουράσω, όμως ε, εγώ θεωρώ ότι έχει πέντε σημεία εύθραστης κατάστασης η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι ένα από αυτά είναι το ότι λείπει μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο σχέσεων με τις τρίτες χώρες, γι' αυτό η έκθεση αυτή αναφέρει και το νέο πλαίσιο σύνδεσης με τις τρίτες χώρες, το λεγόμενο σύμφωνο, το Compact και θέλουμε εδώ να διευρύνουμε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει πραγματικά κίνητρα αυτό δεν θα ήταν παρά η αρχή μια κατάλληλη απάντηση. Σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερα μέτρα μακροπρόθεσμα, ιδίω αντιμετωπίζοντας τις κύριες αιτίες της αναγκαστικής μετακίνησης μέσω της διασφάλισης της ειρήνης της δημοκρατίας και της ασφάλειας, της μείωσης της φτώχειας και της ανισότητας, της ενίσχυσης των βασικών υπηρεσιών, της καταπολέμησης των αδυναμιών των κρατών και της πρόθεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πρόθεσης της καλής κυβέρνησης. Η έκθεση επίσης εκφράζει την, την ανησυχία της για τη σύραξη στη Συρία και φυσικά εμείς υποστηρίζουμε το Λίβανο και την Ιορδανία που συνεχίζουν να δείχνουν μια εξαιρετική αλληλεγγύη φιλοξενώντας χιλιάδες άτομα και δείχνουν μια αλληλεγγύη που είναι δυσανάλογη με την πραγματική τους οικονομική ικανότητα καθώς έχουν περιορισμένους πόρους οι δύο αυτές χώρες. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω ήδη, Πρόεδρε, για να δώσω τη δυνατότητα στους, στους συναδέλφους να τοποθετηθούν απέναντι στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τους συνεισηγητές. Εννέα ομιλητές ζήτησαν το λόγο. 11.30 πρέπει να τελειώσουμε για να κάνουμε την ψηφοφορία για το βραβείο Ζαχάροφ. Θα είναι σύντομες ή παρεμβάσεις ενάμιση λεπτό ο καθένας. Ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματικότητα ότι όπως είπε η κυρία Βαλενθιάνο είναι μια έκθεση πρωτοβουλία. Δεν πρόκειται με μια έκθεση πρωτοβουλία να αλλάξουμε τόσα πολλά πράγματα τα οποία έχουν γίνει με λαθασμένο τρόπο, τις λαθασμένες προσεγγίσεις που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική της και ιδίως τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης των προσφύγων και την κρίση της μετανάστευσης. Παρ' όλα αυτά αυτή η έκθεση είναι ένα καλό εργαλείο για να μπορέσουμε να εκφράσουμε και πάλι την άποψη του Κοινοβουλίου και να εκφράσουμε την διαφωνία μας με ορισμένες από τις ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες ή και τα τελευταία χρόνια. Η έκθεση αυτή λοιπόν ακολουθεί τη γραμμή αυτή που έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το να παρουσιάσει προτάσεις, προτάσεις που έχουν σε μεγάλο βαθμό γίνει δεκτές και από την Κομισιόν, αλλά τα κράτη-μέλη δεν τις έχουν εφαρμόσει. Αν τα κράτη-μέλη είχαν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους στα διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια που ασχολήθηκαν με τα θέματα των μεταναστών που φτάνουν στα σύνορά μας και τις ακτές μας, Εάν είχε υπάρξει <clears throat> μία επανεγκατάσταση των ε, προσφύγων, η ευρωπαϊκή κοινωνία θα είχε δεχτεί πολύ καλύτερα τα μέτρα αυτά, γιατί είναι πολλοί, δήμοι στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν και πόλεις που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Στα Ηνωμένα Έθνη συζητήθηκε πριν από λίγε εβδομάδε το θέμα αυτό και αυτή τη στιγμή επαρχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μονάχα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι παγκόσμιο πρόβλημα, είναι πλανητικό πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε <clears throat> ότι πριν από την κρίση προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχαν δεκάδες εκατομμυρίων εκτοπισμένων ατόμων στον κόσμο ως αποτέλεσμα πολεμικών ενεργειών, ως αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών. Ότι δεν υπήρχαν τέτοιες μεγάλες μετακινήσεις ανθρώπων που θέλουν να ξεφύγουν όχι μόνο από τον πόλεμο, αλλά πολλές φορές και από την πείνα. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω απόλυτα αυτό το οποίο λέει η έκθεση, ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό πρέπει να είναι μια παγκόσμια ευθύνη στην οποία πρέπει να δώσουμε μια παγκόσμια και μακροχρόνια απάντηση. Συγχρόνως όμως υπάρχει η ειδική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βαθμό που οι χώρες μας είναι και μεγάλοι δωρητές, μεγάλοι χορηγοί. Ξέρω ότι ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Θα ήθελα να πω στον κύριο, είπα στον κύριο Διαστεμέρα μόνο τα, τις που θα καταθέσω. Απλώς και μόνο θέλω να υποστηρίξω ένα σημείο, ότι οι συμφωνίες μας με τρίτες χώρες θα πρέπει να κινούνται μέσα στα πλαίσια του διεθνούς ανθρωπιστικού πλαισίου και η βοήθεια που δίνουμε θα πρέπει να είναι χωρίς όρους. Ο Charles Γκέρνς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε μια κοινή ανάγνωση των μεταναστευτικών ροών. Καταρχήν επιμείνουμε στο γεγονός ότι πέρα από τους πρόσφυγες το 90% των ε, μεταναστευτικών ροών είναι μεταξύ των διαφορών περιφερειών. Στην υποσαχάρη Αφρική μεταστεύουν οι άνθρωποι εντός της ίδιας περιοχής. Από τη μία χώρα στην όλη και μόνο το 10% εγκαταλείπει αυτή την περιοχή, 5% για την Ευρώπη και το υπόλοιπο 5% για την Αμερικανική Ήπειρο. Δεύτερον, ας έχουμε και μια κοινή ανάγνωση της ευρωπαϊκής τάσης απέναντι στο φαινόμενο, γιατί όταν πρόκειται για τους πρόσφυγες όλοι συμφωνούν και λένε πρέπει να σεβαστούμε τις συνθήκες της Γενέβης και όταν ε, ερχόμαστε στα πρακτικά πράγματα, η κυρία Μέρκελ αισθάνεται πάρα πολύ μόνη ως προς την υποδοχή των προσφύγων. Ας ε, έχουμε το κουράγιο να πούμε, ας μοιραστούμε το άχθος. Μπορούμε να το πούμε εκατοντάδες φορές ακόμα, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Στο γεγονό ότι κάποιες χώρες δεν θέλουν κανένα πρόσφυγα, άλλες λένε θέλουμε μόνο χριστιανούς, άλλες λένε δεν θέλουμε καθόλου. Έτσι λοιπόν ε, ουσιαστικά έχει πολύ κακές επιδόσεις η Ευρώπη και εγώ θέλω να αποτύσω φοροτιμή στην κυρία Μέρκελ. Τι πρέπει να κάνουμε. Επίσης πρέπει να αποφύγουμε το εξής. Αν θεωρούμε την ε, αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι μπορεί να κάνει τα πάντα για να χρηματοδοτήσει την ε, κλιματική αλλαγή, τις μεταναστευτικέ ροές, ε, για να παρέμβει παντού σε όλους τους τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μέσα δημοσιονομικά. Αυτό θα είναι το τέλος της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε φαντασία και θα πρέπει να είμαστε αδιάλακτοι σε σχέση με τη διατήρηση και την προστασία των μέσων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την αναπτυξιακή πολιτική από δημοσιονομική σκοπιά. Η δέσμευση ε, που θα έπρεπε να έχουμε ε, ουσιαστικά είναι λοιπόν, πολύ παλιά, λείπει 0,3% αλλά αυτό γιατί, για να αποφύγουμε ένα μέλλον που οι άνθρωποι θα εγκαταλείπουν τις αιστείες τους, την περιοχή τους. Γιατί αφενός ε, επενδύουμε χρήματα στην αναπτυξιακή πολιτική για να καταπολεμήσουμε τις αιτίε, αλλά από την άλλη στερούμε από την πολιτική αυτή τώρα παράγει αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε ό,τι αφορά την υποδοχή των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τις περιφερειές τους και να δώσουμε μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα, να δώσουμε θεωρήσεις πολλαπλή πολλαπλής εισόδου σε ανθρώπους που είναι ήδη καταρτισμένοι, άνθρωποι αυτοί που έρχονται από την Αφρική και, ή από αλλού και ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, δεν θα μείνουν εδώ αιωνίως, ούτε θα είναι σε παρανομία. Σας ευχαριστώ. Αν μπορείτε να σεβαστείτε και το χρονικό όριο θα βοηθήσει. κ. Λούκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δώστε μου λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί 1,5 λεπτό δεν φτάνει για μια τόσο σημαντική έκθεση. Απογοητεύτηκα διαβάζοντας την έκθεση, γιατί νομίζω ότι δεν είναι τίποτε περισσότερο από δήλωση καλών προθέσεων, συλλογή στόχων, που σίγουρα μας βρίσκουν όλους σύμφωνους, έκφραση επιθυμίας για βοήθεια, αλλά η πραγματικότητα στα πλαίσια των οποίων δρούμε ε, παραγωνίζονται. Είναι χαρακτηριστικά λέει στην έκθεση ε, πρέπει να δημιουργηθεί νέο αφήγημα στην μεταναστευτική πολιτική. Πιο θετικό αφήγημα. Ε, το πρόβλημα που διαπιστώνω μεταξύ πολλών πολιτών είναι ότι παραείνε και παραπαρουσιάζεται ως θετικό το αφήγημα, ε, παραγωνίζοντας έτσι το πρόβλημα. Ε, το ίδιο και στην έκθεση. Θα περιοριστώ λόγω χρόνου σε λίγες παρατηρήσεις. Αλλά εδώ δημιουργείται εντύπωση ως εάν μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι μας επιτρέπουν οι περιορισμένοι μας πόροι. Όταν μιλάμε για διαχείριση των προσφύγων, πρέπει να ομολογήσουμε ότι η διαχείριση σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα λέμε και όχι. Ενώ το όχι δεν φαίνεται στην έκθεση αυτή. Δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τον καθένα να ασκήσει τα πλήρη δικαιώματά του ανεξάρτητα από το λόγο της φυγής. Ούτε αυτό είναι αλήθεια δεν είναι η αλήθεια με βάση την πραγματικότητα. Η διαχείριση σημαίνει ότι κάποιες φορές θα πούμε ναι, άλλες όχι. Και το πώς θα πούμε το όχι, πώς θα φυλάσσουμε τα σύνορα, πώς θα διαλέγουμε μεταξύ των διαφορετικών ομάδων προσφύγων, αυτό δεν φαίνεται καθόλου στην έκθεση. Τώρα, για την ανάπτυξη. Να πω ότι πρέπει να γραφτεί στην έκθεση ότι η ανάπτυξη σίγουρα είναι πολύ σημαντική, αλλά η αναπτυξιακή πολιτική δεν θα μας λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ε, είναι σταγόνεν το ωκεανό. Όταν λέμε ότι οι ροές προσφύγων, ιδιαίτερα των μεταναστών, ε, είναι ευθύνη της παγκόσμιας κοινότητας, ε, όταν πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες ε, πρέπει να πω ότι είναι ευθύνη εκείνων των κρατών που δεν ε, μπορούν να εξασφαλίσουν οικονομικές συνθήκες κατάλληλες στους πολίτες τους. Θα πρέπει στις χώρες εκεί να υπάρχουν οι δυνατότητες. Ναι, ξέρω ότι ξεπέρασα το χρόνο. Να προσθέσω και να προσθέσω και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να έχουμε σωστό έλεγχο. Όταν κάνουμε ανθρωπιστική πολιτική που δημιουργεί νέες συνθήκες διαβίωσης, αυτό δημιουργεί και παράγοντες έλξης που θα πρέπει να απασχολήσουν επίσης την έκθεση αυτή. Θα, είναι οι παράγοντες έλξης πολύ μεγάλη. Ξέρω, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε για το Σαχάροφ σήμερα. Έχουμε λίγο χρόνο. Ε, τώρα δεν μπορούμε να αναβάλουμε το επόμενο θέμα. Η κυρία Αλμπιόλ. Ευχαριστώ. Εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω με πολλά πόσα είπε η κυρία Βαλενσιάνο και με κάποια πόσα είπε ο κύριος Δίας Δεμέρα, όμως ε, δυστυχώς όλα αυτά που σχολιάσατε εσείς δεν παρουσιάζονται στην έκθεση. Εγώ νομίζω ότι στην έκθεση αυτή δεν γίνεται η κατάλληλη εστίαση. Καταρχήν, για το πιο βασικά δεν γνωρίζετε το ανθρώπινο δικαίωμα να μεταναστεύσει κανείς και δεύτερον κάθε φορά που μιλάμε ε, ουσιαστικά για τις χώρες προέλευσης δεν προτείνονται λύσεις, ε, ούτε δίνονται θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, ούτε για να τεθούν τέλος σε πολιτικές, ε, στο εμπόριο όπλων που δημιουργούν τις σειράξεις. Αλλά η έκθεση αυτό που κάνει είναι στο να προωθεί περισσότερο την εξορτικοποίηση των συνόρων και να ε, προωθεί τις συμφωνίες αυτές τις ντροπιαστικές όπως είναι η συμφωνία με την Τουρκία ή το Αφγανιστάν. Όταν ε, συνδέεται στην έκθεση η το αφγανισταν οταν συνδεεται στην εκθεση μεταναστευση με την ασφάλεια, τι γίνεται εκ νέου και για μια ακόμη φορά σε αυτό το κοινοβούλιο, ποινικοποιούνται οι μετανάστες. Επίσης, βλέπουμε ότι εδώ επιλέγεται η στρατιωτικοποίηση των συνόρων και μάλιστα στην έκθεση υποστηρίζεται η αποστολή UNAFOR για να στέλνονται, να στέλνονται πλοία από το ΝΑΤΟ για να σταματούν τις βάρκες με τους μετανάστες. Ε, εδώ αναφέρουμε την κλιματική αλλαγή μέχρι την εκμετάλλευση των εργαζομένων ε, και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. αυτό δεν προσοκιστεί ούτε η περικοπή του προπολογισμού για τη συνεργασία. Παραδείγματο χάρη, το Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία έκανε μεγάλες ε, περικοπές ε, και ούτε αναφέρεται αυτό το ζήτημα στην αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης, αυτό που προωθείται είναι να επιστραφεί στην χώρα του οποιοδήποτε έρχεται στην Ευρώπη. Και για τα ΚΑΠ, τα μία ταμεία, τι γίνεται από τότε που συμφωνία στη Βαλέτα να χρηματοδοτούνται και να εξοπλίζονται ε, δυνάμεις σε χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ούτε βρίσκουμε κάτι τέτοιο στην έκθεση. Και τελειώνω γιατί θα παρουσιάσουμε και τις κατάλληλες ε, τροπολογίες. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται λόγος για αυτό που εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να λέγεται στην έκθεση Τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να φύγονται αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κοιτάω συνέχεια το ρολόι, μιλώ και με τον κύριο Μπρόκ εδώ. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε όλους και να κάνουμε συζήτηση σωστή. Λοιπόν, οι δύο συνεισηγητές τι λένε, να τελειώσουμε τώρα και να προγραμματίσουμε κι άλλη συνάντηση γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να πούμε πολλοί συνάδελφοι, αλλά η ψηφοφορία για το βραβείο Σακάροφ πρέπει να αρχίσει στις 11.30. μπορεί να είναι και δύο γύροι ψηφοφορίας, είναι, είναι επίγον. Να βρούμε ο κύριος Μπροκ και εγώ κάποιο χρόνο για να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή που δεν πρέπει να την κλείσουμε άρον-άρον. Είναι πολύ σημαντική. Ε, η ομάδα των Πρασίνων δεν μίλησε. Δύο σκιώδεις εκεί. Λοχ Μπίλερ και Χάουταλα. Ποιος θέλει να μιλήσει. Και οι δυο να μιλήσουν και να πάρουν από ένα λεπτό. Η κυρία Λοχ Μπίλερ. Ωραία. Και η άλλη συζήτηση θα γίνει αργότερα. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε βέβαια με πολλά ουσιαστικά θέματα της έκθεσης. Πιέζει ο χρόνος όμως να πω ε, την κριτική. Υπάρχει έκθεση άφετ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση στις τρίτες χώρες και συγκρίνουμε ε, την έκθεση αυτή και τις, ε, τα εκτιμώντας και τις αιτιολογικές σκέψεις και είναι επικάλυψη σχεδόν 100%. Οι δύο εισηγητές να το σκεφτούν αυτό. Και η κυρία Βαλενσιάνο πρέπει να είναι πιο σαφής όταν είπε στην αρχή ότι υπάρχουν τόσε τροπολογίε που κάνατε παράλληλη έκθεση. Τι σημαίνει αυτό για τις διάφορες τροπολογίες. Επίσης, για την ε, διαμεσολάβηση, την ε, πρόληψη των συγκρούσεων, τα αίτια και τις ρίζες των προβλημάτων, τις ε, βίες συγκρούσεις, αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε καλύτερα. Επίσης, για την διαδικασία του χαρτούμ δεν λέτε τίποτα, γιατί γίνεται μια πολύ σοβαρή προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την κυβέρνηση του Σουδάν για να βρεθούν τρόποι, πώς να το πούμε, να μείνουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα είπα έτσι πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ε, ένας από κάθε ομάδα έχει οριστεί, αλλά δεν θα προλάβουμε. Δεν λυπάμαι πάρα πολύ. Περισσότερες, ε, περισσότερες σκιώδες από διάφορες ομάδες δεν μίλησαν, αλλά δεν φτάνει ο χρόνος, έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον μια ώρα, μια ώρα και ένα τέταρτο, για να προλάβουμε να τα πούμε όλα και οι σκιώδεις. Θα το αναβάλουμε. Δεν θα μπορέσω να δώσω το λόγο σε άλλους. Δεν ξέρω αν οι δύο εισηγητές, ένα λεπτό καθένας, οι δύο εισηγήτριες, οι δύο εισηγητές ε, και μετά θα σας δώσω το λόγο όταν θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Προηγείται το αγώ. Μονάχα να τονίσω την ιδέα ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στη συζήτηση όπως είπε και η Πρόεδρος και στη συνέχεια εμείς θα εξετάσουμε τις τροπολογίες που καταθέτουν οι ομάδες. Αυτή είναι μια πολύπλοκη έκθεση αλλά φυσικά δεν μπορεί να τα καλύψει όλα. Είναι πολλά πράγματα που δυστυχώ δεν χωράνε στην έκθεση. Η θέλησή μα είναι βέβαια να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απόψει από αυτές που έχουν διατυπωθεί εδώ σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο κύριο ε, Ντιεμέρα. Και εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η Ελένα. Θα λάβουμε υπόψη ιδιαίτερα αυτά που είπε ο Ερή, Λούκε, Καμπιόν, Αλιβιόρ και μια στιγμή. Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ξέρω ότι ήρθατε να ψηφίσετε, αλλά παρακαλώ αφήστε τον εισηγητή μας να μιλήσει. Παρακαλώ να σιωπήσετε και να κάνετε ησυχία. Ο Αγουστίν και πάλι. Ναι, έλεγα ότι σίγουρα η κυρία Χάουταλα ξέρει πόσο εκτιμώ τις ιδέες της, που είναι πάντα επικοδομητικές. Σας υπενθυμίζω όμως ότι η διαδικασία του Χαρτούμ αναφέρεται στο σημείο 14 της έκθεσής μας. Αυτά λοιπόν και θα συνεχίσουμε να συζητούμε το θέμα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, ναι, δεν είχαμε αρκετό χρόνο για αυτή τη συζήτηση, ώστε να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο. Η Ελένα και ο Αγουστίν θα πρέπει να σας ρωτώ να κρατήσουμε την προθεσμία για τις τροπολογίες 18 Οκτωβρίου. Εάν ναι, θα έχουμε μια περαιτέρω συζήτηση με τις τροπολογίες πριν ψηφίσουμε, δεν ξέρω αν αυτό θα καθυστερήσει την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Θα έχουμε λοιπόν και μια νέα κοινή συζήτηση των δύο επιτροπών με τις τροπολογίες πια και θα έχουμε μια καλύτερη ιδέα για το τι θέλουν οι συνάδελφοι στο θέμα αυτό. Η προθεσμία τροπολογιών λοιπόν είναι 18 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Η επόμενη τρίτη το μεσημέρι λοιπόν και ξανα, θα ξαναδώσουμε τότε τη δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να μιλήσω για το θέμα αυτό. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο τώρα, τον κύριο Μπροκ, αλλά σας παρακαλώ σταματήστε τα πηγαδάκια εδώ στα δεξιά μου. Ο κύριος Μπροκ θα είναι πιο στεναρός στο να του ζητήσει να κάνει ησυχία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Έλμαρ. Νομίζω ότι αυτή η άσκηση μεταξύ των δύο εισηγητών να προσπαθήσουμε να φέρουν πιο κοντά τις απόψεις τους, κάτι που γίνεται και στην Ισπανία. Κυρίες και κύριοι, είναι και κλεισμένο των θυρών η, συνάντηση, η συζήτηση αυτή. Παρακαλώ όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα να είναι εδώ να αποχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό και σταματήστε τα πηγαδάκια σας παρακαλώ. Είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Ja, das muss der Frau nehmen, der muss ich gleich reden.